Ντελούκα για τα θέματα μέρη μα και επιμέλεια. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Είμαι εγώ η Πατρίτσια Ντελούκα και θα σα μιλήσω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικώ και κατόπιν να δώσω τη σκητάλη στου άλλου συναδέλφου για τα πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτα, πρώτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να εκφράσει την αλληλεγγύη της ε, προς ε, όλα τα θύματα απαγωγής των ανηλίκων, διεσμένων διακρίσεων, βίες συμπεριφοράς προς τους ε, γονείς επίσης που δεν τους επιτρέπεται να έχουν επαφή με τα παιδιά τους. Ακούσαμε κάποιες περιπτώσεις ε, τις οποίες ε, ήδη ε, μας έχουν απασχολήσει και ήδη έχουμε διαβιβάσει έγγραφος απαντήσεις. Και ευχαριστούμε τους υποβάλλοντες την αναφορά που μας ε, ενημερώνουν για την εξέλιξη αλλά πάντως ε, θα σας πω ότι ο πλευράς νομικής για αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει αλλάξει η κατάσταση και είπαμε και τα ίδια σε μια προηγούμενη συνέντευξη μας το 2013 εδώ έχουμε κάποιες νέες αναφορές κάποιες άλλες που στο μεταξύ έχουν υποβληθεί και εγγράφους. Λάβαμε μόλις χθες ε, για κάποιες από αυτές τις αναφορές στην ε, τεκμηρίωση και πρόκειται για περιπτώσεις που όπως γνωρίζετε αφορούν πολύ μεγάλη ποικιλία καταστάσεων. Μιλούμε για απαγωγή, προβλήματα με τη γονική με την επιμέλεια, το δικαίωμα επισκέψεως, ε, την ε, βία στην οικογένεια, ε, την καταπάση θεμελών δικαιωμάτων, δυσμενείς διακρίσεις λόγω ηθαγενείας, αλλά και ακόμα και παραμέληση της παροχής ιατρικής βοήθειας ή η απαγόρευση προσβασιμότητας σε έγγραφα. Όλα, αλλά όπως και στο παρελθόν να σας δώσουμε μια γενική εποπτεία του πώς έχει η κατάσταση πώς έχει η κατάσταση τι, τι, τι διέπει πλευράς νόμου στις περιπτώσεις αυτές. Επί της αρχής μιλούμε για πράξεις και παραλήψεις κατών μελών επ' αυτού έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου και σε σχέση με τον έλεγχο από πλευράς Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για τις περιπτώσεις που σήμερα εξηγήθηκαν, από ό,τι φαίνεται, η περίπτωση δεν καλύπτεται από το κοινωτικό δίκαιο. Συγκεκριμένα τώρα. Το πώς έχουν κρίνει κάποιες αυτές τις υποθέσεις οι δικαστικές αρχές ή το πώς λειτουργούν οι υπηρεσίε κοινωνικής πρόνοιας στη Δανία. Επίσης, η Δανία διέπεται από ειδικό καθεστώς δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. εξαιρείται η χώρα της εφαρμογής των όσων διέπουν τις υπόλοιπες χώρες από πλευράς ε, χώρου, ενίου χώρου δικαιοσύνης, ελευθερίας κλπ. Οπότε έχουμε έναν κανονισμό σε σχέση με την ευθύνη των γονέων ο οποίος ούτε αυτός εφαρμόζεται στην Δανία, που ξέρετε τις εφαρμογές του δηλαδή. Ίσως έχουμε κάποιες άλλες διεθνείς ε, συμφωνίες που μπορεί να ισχύουν, όπως ας πούμε η Διεθνή Σύμβαση για την ε, Απαγωγή Ενηλίκων. Είναι σημαντικό πάντως να τονίσουμε ότι το κοινοτικό δίκαιο ρυθμίζει μόνο τα ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή, εάν έχει αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση το δικαίωμα επίσκεψη σε ένα κράτο μέλο, μπορεί ο γονέα να επιδείξει την αναγνώριση τη απόφαση σε άλλο κράτο αλλά όμω επί τη ουσία δεν μπορεί να κρίνουμε. Παραμένει αυτό εθνική αρμοδιότητα δηλαδή. Συνέπεια τούτου είναι το ότι δεν έχει γενική αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορεί να επισέλθει στην ουσία των καθέκαστων υποθέσεων. Τα συντρέχει περί της φορμής κοινωτικού δικαίου. Και τώρα να δώσω τη σκητάλια στους συναδέλφους. Στην ε, Κλάουδια πρώτα-πρώτα για να σας εξηγήσει τι ισχύει όσον αφορά την βία στην οικογένεια και την προστασία των θυμάτων. Uh, yes, thank you. Ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο, δύσκολα αυτά που ακούμε. Εγώ συγκινήθηκα από όλα όσα άκουσα σήμερα. Παρόλα αυτά, ως Κομισιόν, πρέπει φυσικά να απαντήσουμε πιο επίσημα. Η μονάδα μου ασχολείται με το ποινικό δίκαιο, γι' αυτό, για αυτές τις πτυχές θα μιλήσω για την προστασία θυμάτων εγκληματικής βίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει την κατάσταση των θυμάτων εγκλημάτων στην Ένωση και αυτό συμπεριλαμβάνει βέβαια και τα θύματα οικιακής βίας καθώς και σεξουαλικής παρενόχλησης Υπάρχουν δύο σημαντικά εργαλεία. Υπάρχει η οδηγία του 12 που βελτιώνει τις διαδικασίες εφαρμογής των δικαιωμάτων, άσκησης των δικαιωμάτων των θυμάτων και η οποία βοηθάει πραγματικά τα θύματα να προστατευθούν κατά τις ποινικέ διαδικασίες, να προστατεύονται, να πληροφορούνται και υπάρχει και ένα άλλο εργαλείο που αφορά τα θύματα για τα μέτρα προστασίας θυμάτων όταν βγαίνουν από τη χώρα προέλευσής τους. Συμφωνώ βέβαια με αυτά που ήδη είπε η συνάδελφός μου η Δανία, ε, αντιμετωπίζει ιδιαίτερη κατάσταση ως προς την εφαρμογή όλων αυτών των νομοθετημάτων γιατί δεν δεσμεύεται ούτε από την οδηγία του 12 η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται βέβαια μόνο το 15 αλλά ούτε τότε θα δεσμεύεται η Δανία. Δεν υπάρχει λοιπόν ενωσιακός νόμος στη Δανία για αυτά τα θέματα. Και το ίδιο ισχύει και για τα δύο άλλα νομικά εργαλεία, την προστασία σε περίπτωση που κάποιο θύμα φεύγει από τη χώρα προέλευσης του πάλι δεν δεσμεύεται η Δανία και άρα δυστυχώς μόνο αυτό μπορούμε επίσημα να απαντήσουμε ότι δεν έχουμε δικαιοδοσία παρέμβασης στη Δανία. Ευχαριστούμε για αυτήν την απογοητευτικότατη για αυτό το απογοητευτικότατο συμπέρασμα τίποτε άλλο ναι ο επόμενος η επόμενη ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε εγώ εργάζομαι με τον συντονιστή των δικαιωμάτων των παιδών στην Κομισιόν. Να σας πω μερικά για αυτό που κάνουμε και που αφορά λιγάκι αυτά που είπατε σήμερα. Πρέπει να τονίσω ότι αυτά όμως είναι από την πτυχή της γενικότερης πολιτικής και όχι των συγκεκριμένων αναφορών που ακούσαμε σήμερα. Πρώτον, κάτι στο οποίο συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζήτησε από την Κομισιόν να επεξεργαστεί ένα πιλωτικό επιραματικό σχέδιο για την πληροφόρηση των ζευγαριών σχετικά με την γονική ευθύνη σε περίπτωση χωρισμού ή διαζυγίου. Είναι σημαντικό να έχουν τη σωστή πληροφόρηση όλοι για την περίπτωση που θα προκύψει κάποιο πρόβλημα σε ζευγάρια διαφορετικών εθνικότητων. Δεν είναι συγκεκριμένη νομοθεσία ούτε μελέτη, είναι απλώς ένα πρόγραμμα πληροφόρησης. Δεύτερον, υπάρχει μια, αναλάβαμε μια μελέτη για τα παιδιά που εμπλέκονται σε δικαστικές διαδικασίες και που αφορά όλες τις χώρες μέλη αφορά ποινικέ διαδικασίες και αστικές διαδικασίες αλλά και θέματα που αφορούν δικαιώματα μέρημνας και επίσκεψης κλπ. Λοιπόν, προ αυτή τη φορά πρόκειται για μελέτη. Θέλουμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού και πώς εφαρμόζονται οι διαφορετικές νομοθεσίες στις χώρες μέλη για να βγάλουμε συμπεράσματα. Τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ότι επεξεργαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των παιδών στις χώρες μέλη. Και για να είμαστε σαφείς, η Ένωση καθεαυτήν δεν έχει δικαιοδοσία για τα εθνικά συστήματα προστασίας των παιδών. Η ιδέα είναι απλώς να οθήσουμε τα κράτη-μέλη, να τα βοηθήσουμε να δουν τα πράγματα πιο ολοκληρωμένα, πιο σφαιρικά, γιατί συχνά τα παιδιά και γονείς καμιά φορά εμπλέκονται σε καταστάσεις που δεν αφορούν μία μόνο διάσταση, αλλά διάφορες μαζί. Διάφορους θεσμούς, πρακτορία, υπηρεσίες των χωρών μελών ή και πολλές χώρες μέλη. Προσπαθούμε λοιπόν πάλι να καταγράψουμε τα πράγματα, να τα χαρτογραφήσουμε, να δούμε τι ισχύει στα διάφορα συστήματα προστασίας των παιδών στις χώρες μέλη για να μπορέσουμε τελικά να συγγράψουμε, να συντάξουμε κατευθυντήριες γραμμές. Πώς θα μπορούσαν ας πούμε οι γονείς να χρησιμοποιήσουν χρηματοδότηση κτλ. Ευχαριστούμε. Δεν θέλει άλλος από την Επιτροπή το λόγο. Λέει η Πρόεδρος. Άρα Ο κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί αναφερόμενοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για μια από αυτέ τι οδυνηρέ μέρε που μα μένουν στο μυαλό γιατί, γιατί, γιατί βλέπουμε τα όρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όρια του οράματό μα και βλέπουμε αυτή την συμπεριφορά που προέρχονται από τι ε, αρχέ κάποιου κράτου μέλου. Οπότε και Βέβαια, πρέπει να λάβουμε δράση και ευθύ εξ αρχή ήξερα από την αρχή της πολιτική μου θεωρημίας ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγη μπήκαν για να μετρηθεί, να αξιολογηθεί η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών μιας υποψήφιας χώρας. Ουδέποτε όμως δεν φαντάστηκα ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης κάποια στιγμή θα ε, ισχύαν σε σχέση με μια τέτοια κατάφορη παραβίαση των δημιουργικών δικαιωμάτων. Είναι πραγματικά απίστευτο. Λατρεύω τη Δανία και ανέκαθεν έτρεφα μεγάλη εκτίμηση για την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα εκείνη. Αλλά όταν ακούω κυρίω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και αυτέ τι ε, τραγικές καταθέσεις των αναφερομένων ε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία ε, θα πρέπει να σας απασχολήσουν ε, κύριοι τη Επιτροπή. πρωτα Πρώτα-πρώτα, τι απέγινε η ίση μεταχείριση των γονείων ενώπιον τη δικαιοσύνης. Είναι το βασικό δικαίωμα τη ίση μεταχείριση ενώπιον τη δικαιοσύνης που ισχύει για του Ευρωπαίου πολίτες. Εδώ διαπιστώνεται κατάφορη δυσμενής διάκριση σε σχέση με την ηθαγένεια, με την εθνοτική καταγωγή, σε σχέση με το ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκή Ένωση δεν απολάβουν η συμπαχείριση από τη δικαιοσύνη, από τις κρατικές αρχές. Αυτό, αυτό αντιβαίνει στο κοινοτικό δίκαιο. Στην δύστιχη την Ρουμανία, στη φτωχή Ρουμανία, εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια μεταχείριση, θα ήμουν ο πρώτος που θα ζητούσε την τιμωρία της χώρας, διότι είναι απλώς απαράδεκτο. Αυτό αντιβαίνει στα οικονομικά δικαιώματα των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνταχείριση των διαδίκων. Κάτι το οποίο δεν ίσχυσε, σύμφωνα με όσα μας λένε οι αναφερόμενοι. Πάντοτε μόνο η μία πλευρά είναι η προνομιούχος. Η άλλη πλευρά, ο άλλος διάδικος, αποστερείται των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Και δεν μιλάμε για τη Ρωσία ή άλλες χώρες, μιλάμε για ένα κράτος μέλος της Ένωσης. Επίσης, πρόκειται για την απόφαση των στομικών αρχών να κρατήσουν, να κατακρατήσουν αφαιρώντας το διαβατήριο ενός ε, πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταπατώντας ε, το θεμελιώδες δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Ακόμα και σε μη κρατημένη απόφαση του να κρατήσει ε, κάποια αρχή το διαβατήριο και έτσι να περιοριστεί η δυνατότητα διαμονής και διακίνησης, αυτό απαιτεί δικαστική απόφαση. Εδώ μιλούμε για απόφαση της αστυνομίας. Αυτό δεν είναι αστυνομική αρμοδιότητα. Γιατί επειδή είναι αστυνομία τη πρόκειται για κάτι απαράδεκτο. Πρόκειται για βίαιη επέμβαση των ε, κρατικών αρχών στην ε, οικογένεια, στις σχέσεις παιδιών και γονέων, στη Σπάρτη. Υπήρχε ο δρακόντιος νόμος, αποφασιζόταν ποιο παιδί είναι εντάξει και ποιο δεν είναι. Όταν υπήρχε δηλαδή κάποια αναπηρία καταδικαζόταν το παιδί σε θάνατο. Μα είναι δυνατόν να αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάποια αρχή να αποφασίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό για μια οικογένεια. Είναι κατακλείδη. Είναι Παράδειγμα αυτό να γίνεται έτσι μόνο πλευρά. Με σοκάρει. Νιώθω τόσο στεναχωρημένος. Είναι τόσο δυνηρό αυτό το να ακούμε αυτές τις απίστευτες ιστορίες. Επίσης, πώς είναι να μια αρχή οπουδήποτε να αποστερεί το θεμελιώδης δικαίωμα του γονέα να έχει πρόσβαση, να δει, να επισκεφτεί το παιδί του ή το παιδί της. Πώς θα τον ένας ε, γονέας να φυλακίζεται. Δεν έχει σημασία μία μέρα ή ένα χρόνο. Απλώς και μόνο διότι προσπάθησε να έρθει σε επαφή με το παιδί του ή το παιδί της. Τι είναι αυτό, αυτό είναι σε ένα ναζιστικό καθεστώς το οποίο αποφασίζει για το πώς θα ρυθμίσει την οικογενική ζωή, τη σεξουαλική ζωή, το τι γίνεται με τα, με τα παιδιά. Είναι δυνατόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο έτσι με τόση αφέλεια. Λυπάμαι, λυπάμαι που μιλώ με τόση σκληρότητα, αλλά και εγώ είμαι γονιός. Το παιδί μου πέθανε από λευκαιμία. Έχω τώρα μια, ένα ανιψιό. Ξέρω τι πάνε Πώ είναι δυνατόν κάποιος να αποφασίζει με τέτοιο ε, τρόπο οριστικό για τα δικαιώματα ενό γονιού. Συγγνώμη, αλλά αυτό με σοκάρει. Συμπαθάτε μου. Κύριος Ποστινάρο συνεχίζει. Παρακαλώ συγχωρήστε με για αυτή την τόσο έντονη συναισθηματική φόρτιση και αυτά τα οποία σας είπα. Αυτό δεν είναι το να συνεχιστεί έτσι. Απλώ δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν έτσι. Δεν είναι business as usual. Δεν είναι θέματα ρουτίνα. Δεν συζητούμε τώρα για εμπορεύματα, για εμπορικά δικαιώματα, για, για πνευματική ιδιοκτησία. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Άρα ας έχουν τουλάχιστον κάποια κοινά στάνταρ, κοινά πρότυπα για τα παιδιά και τους γονείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την μεταχείρισή τους. Μα ή το να κατεβαίνουμε στον κόσμο και να λέμε για την προλογική εκστρατεία τι ωραία, τι απίστευτα όμορφο είναι το ευρωπαϊκό όραμα. Και τι θα πούμε στους αναφερόμενους, τι θα πούμε στους άλλους γονείς στην Ευρώπη που μας είπαν, να ακούσαμε τι γίνεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι μήνυμα να τους δώσουμε αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι να πούμε στους ανθρώπους αυτούς, τι απάντηση να τους δώσουμε. μην αναμένουμε σιωπή, να σιωπούμε ενώπιον αυτών. Άρα, ουδετερότητα εδώ σημαίνει συνενοχή. Εδώ θα βάλω τελεία, πάλι συγχωρήστε με, αλλά όταν μιλούμε για δικαιώματα των παιδιών, δικαιώματα των ελίκων, κανείς δεν μπορεί να είναι ψυχρός και ψύχρεμος και ατσάλινος. Πρόκειται για τα πιο πολύτιμα συναισθήματα. Ακόμα και τα ζώα μεταχειρίζονται τα νεογνά oh, τέλος πάντων. Θα έλεγα ανθρώπινα, με ανθρωπιά. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ψυχροί και ψυχροί όταν μιλούμε τα δικαιώματα των Αγγλικών και να αποδεχόμεθα το να συνεχίζεται μια τέτοια κατάσταση. Θα έλεγα να προτρέψουμε τους αναφερομένους να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά, αλλά, πόσο καιρό θα καταδικαστεί ένα παιδί να μην μπορεί να δει το μπαμπά του ή τη μαμά του, να στερείται του γονιού του έως ότου κρίνει το δικαστήριο του Στρασβούργου. Οπότε το κράτος μέλος μετά να υποχρεωθεί να εφαρμόσει τη σχετική απόφαση. Πώς, πώς να το μετρήσουμε. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι άλλοι λοιπόν. Ερτουγκάι. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Όταν πήγαμε, η Άντζελα, ο Πίτερ και εγώ σε εκείνη την ερευνητική του επιτροπή στην Δανία, τότε αντιμετωπίσαμε κάτι πάρα πολύ ασυνήθιστο, όπω είπε και ο Βίκτορ. Άκουσα τον συνάδελφο και φίλο Μποστινάρο. Είπε για τις προσωπικές του εμπειρίες, το προσωπικό του δράμα. Οπότε δύσκολα τώρα να περιοριστούμε σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Βίκτορ, αυτό είναι μια λεπτομέρεια του όλου τοπίου που αντιμετωπίσαμε τότε στην Δανία. Τι ακούσαμε τότε από, από μητέρες, από έναν πατέρα, το τι περνάνε. Εκεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόκειται για μια τραγωδία. Ότι αυτά γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για κάποια χώρα κάπου μακριά στη μέση της ε, Αφρικής, στα βάθη της Νοτιού Αμερικής. Πρόκειται για κάτι που γίνεται εδώ στην ένωσή μας. Για μανάδες που είναι στριμωγμένες από τέτοιες διαδικασίες, φυλακισμένες, για παιδιά με ψυχολογικά ε, προβλήματα, παιδιά που, που τα έχουν ξεριζώσει από την οικογένειά τους και πρόκειται για παραβιάσει που γίνονται από πλευρά τη Δανία. για τα ανθρωπινά δικαιώματα, για διεθνεί συμφωνίε. Μερικοί αυτό το θεωρούν προοδευτικό. Αυτό γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλη μια φορά, εδώ, θέλω να σας πω κάτι για την ουσία. Άκουσαμε τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας εξήγησαν, είναι αλληλέγγυοι, αλλά Πάντα υπάρχει ένα όμως. Το ε, όμως είναι η επικουρικότητα το ένα το άλλο. Μα αυτό είναι το πρόβλημα αγαπητοί σύντροφοι, συνάδελφοι και φίλοι. Ακούσαμε αυτές τις μανάδες. Τις ξεπετάξαμε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Και μα συγκλώνησαν, μας συγκίνησαν και συνεχίζουμε τη δουλειά σαν να σημαίνει τίποτα. Ε, δεν είναι δυνατόν αυτό να μείνει έτσι εδώ, μέσα σε, αυτό, σε αυτή την αίθουσα, αυτό θα πρέπει να το βγάλουμε πιο έξω. Αυτό θα πρέπει να κατέβει στην Ολομέλεια για να τα ακούσουν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο είναι ένα σκάνδαλο. Γίνεται στην Ευρώπη. Σκάνδαλο της Ευρώπης. Δεν ξέρω ποιο τρόπο θα το χειριστούμε, αλλά είναι από τα πιο σημαντικά που θα πρέπει να αναλάβει κατά αυτή τη θητεία η Επιτροπή μας. Τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ καλή η πρότασή σας, κύριε Τουρκαής. Κύριε Μπουλό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να προσφέρω την ε, συλλογική υποστήριξη προς τους αναφερόμενους, τις αναφερόμενες, με τις τραγωδίες που μας περιέγραψαν, τις τραγωδίες που ζούνε και να τους βεβαιώσουμε ότι όλα τα θέματα που μας απασχολούν εδώ στην Επιτροπή των Αναφορών είναι πάντοτε τα θέματα τα πιο καυτά, τα πιο τραγικά, τα πιο σημαντικά που έρχονται και συζητούμε μέσα στην αίθουσα της Επιτροπής των Αναφορών. Και το λέω αυτό ότι τα συζητούμε με πολύ ταπεινοφροσύνη γιατί ε, μπορούμε να βοηθήσουμε ίσως και να εξασφαλίσουμε την αντιμετώπιση προβλημάτων πολλών των αναφερομένων σε άλλα πεδία περισσότερο από ό,τι στο δικό μας. Ε, όταν λοιπόν ε, δεν υπάρχει οικογενειακή, ε, οικογενειακό κύτταρο, δεν υπάρχει ζωή στην κοινωνία και χωρίς ζωή στην κοινωνία δεν μπορεί κανείς να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος και ως προσωπικότητα. Εμείς δεχθήκαμε αυτές τις αναφορές, θεωρήσαμε παραδεκτές δηλαδή. Για να είναι παραδεκτή μια αναφορή, αναφορά πρέπει να εγγράφεται στο πεδίο των αρμοδίτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι, είναι ευρωπαϊκό το θέμα, δεν ε, αφορά μόνο την επικουρικότητα και ότι υπάρχουν κάποιες πτυχές επικουρικότητας, το αμφισβητώ αυτό. Επίσης δεν ε, πρόκειται εδώ περί επιθέσεως εις βάρος ενός κράτους, έστω και αν η Δανία μπαίνοντα στο ευρωπαϊκό εστιατόριο παίρνει μενού à la carte και ως εκ τούτου θα ήταν εύκολο να προσπαθούσαμε να την πιέσουμε να, να παίρνει το πιο μαζικό μενού και να καταναλώνει πιο μαζικά. Αλλά πάντως δεν είναι μεμονωμένες αυτές ε, οι περιπτώσεις. Είδαμε και στην περίπτωση της Γερμανίας ε, τόσα προβλήματα με εκατοντάδες αναφορές πάνω στο ίδιο ζήτημα και τώρα πάλι βλέπουμε τόσες πολλές αναφορές σχετικές με τη Δανία στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό θα πω στους αναφερόμενους, ότι δεν είναι μόνος του αυτή την υπόθεση, όσο και αν είναι περίπλοκα τα χαρακτηριστικά της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις εδώ στην Επιτροπή των Αναφορών και να ασκήσουμε στο βαθμό που μπορούμε πιέσεις και να βρούμε και εφάνταστες ακόμη λύσεις. Και πρέπει να πω επίσης ότι αυτό είναι η κορφή μόνο του παγόβουνου. Πολλοί είναι οι πολίτε που αντιμετωπίζουν εξίσου σημαντικά προβλήματα και τα ίδια ακόμη, αλλά μη γνωρίζοντα ότι υπάρχει Επιτροπή των Αναφορών, δεν έχουν ε, προσφύγει σε εμά. Έτσι λοιπόν, τα θέματα τη επιμέλεια ε, τέκνων και στη Γερμανία τα έχουμε δει ήδη. Τρία χρόνια τώρα που έχουμε ενασχοληθεί με το θέμα αυτό δεν έχουμε δει προέοδο, θα συμφωνήσετε μαζί μου, Δυστυχώ, Έχουμε κάνει προτάσει, έχουμε επισκεφθεί τη Γερμανία, όπω άλλωστε και με την ε, Δανία. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχει αφαίρεση επιμέλειας δικαιώματος επικοινωνίας με τα παιδιά, προβλήματα ως προς τις διοικητικές ε, διατυπώσεις, δύσκολες διατυπώσεις χρονοβόρες που μερικές φορές το παιδί φτάνει να ενηλικιώνεται και έτσι πλέον δεν έχει και λόγο ύπαρξη διαδικασίας, ε, οι διαδικασίες, κατηγορίες εφάνταστες και παλαβές μέχρι και για απαγωγή παιδών χρήση ακόμη και καταχρηστικά του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, Συλλήψης και Φυλακίσεις και σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω ρωτήσει και από τη Γερμανία να μου απαντήσουν και που αφορούν θέματα που μας έχουν απασχολήσει και σήμερα, ε, λίγο πολύ έχουν να κάνουν με το κοινοτικό δίκαιο και τις αποφάσεις στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και την επικουρικότητα και αντίστοιχα την ομολογία των κρατών μελών. Πρέπει όμως να μην λησμονούμε ότι πολλές φορές η νομοθεσία στα κράτη-μέλη όταν έχουμε μεικτό ζευγάρι μπορεί να είναι αντιφατική από το ένα κράτος στο άλλο και να λαμβάνει η δικαιοδοσία του ενός κράτους απόφαση αντίθετη με αυτή που έχει λάβει η άλλη ε, δικαιοδοτική αρχή. Άρα τι θα κάνουμε, ποιανού η δικαιοδοσία αναγνωρίζεται και επικρατεί. Βέβαια είναι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά το αναγνωρίζω, τα δικαστήρια, τα ε, οικογενειακά δικαστήρια ή το Jugendamt προκειμένου για τη Γερμανία που έχει κάνει καλή δουλειά. Ε, παρ' όλα αυτά μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρεκτροπές και προβλήματα. Και πρέπει κάθε κράτος μέλος να είναι σε θέση να προτείνει στον πολίτη του τη δυνατότητα προσφυγής, πραγματικής προσφυγής, πραγματικού ένδικου μέσου, να μην περνάει δηλαδή από, τον ίδιο, ε, από την ίδια αρχή για να βρει το δίκαιο του. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Σύμβαση Ρώμη 3, η οποία λέει στους πολίτες όταν πρόκειται να παντρευτούν, χωρίς να είναι και πολύ γκλάμουρο όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει τους επισημαίνει ότι υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει ότι σε ενδεχόμενο διαζύγιο μπορούν να υπαχθούν σε αυτή. Αλλά πείτε μου, ποιο δήμαρχο, αντιδήμαρχο για του γάμου αρμόδιου, γιατί και εγώ από τη Γαλλία στο πιο μικρό χωριό, αν φανταστούμε, ξέρει ο αντιδήμαρχος θα κάνει το γάμο ότι υπάρχει αυτή η νομοθεσία για να συμβουλέψει το ζευγάρι ή στη Γαλλία ή στη Δανία ή στη Γερμανία. Ποιος επικαλείται αυτές τις διατάξεις της 3. Παίρνουμε τις ωραίες και μεγάλες αποφάσεις, αλλά τελικά κανείς δεν τις εφαρμόζει όταν πρέπει. Και στις προτάσεις που έχω διατυπώσει για το Jugendamt στο παρελθόν, γιατί ναι, μια, ένα λεπτό ξέρω μου μένει. Η Γαλλία και η Γερμανία, είναι, η, η Γερμανία και η Ιταλία είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν αμοιβαίες ε, σχέσεις σε αυτό. Αλλά ε, πρέπει να μπορούν να έχουν διαμεσολαβητή για τα οικογενειακά θέματα οι πολίτες. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να έχουν κάποιον ο οποίος θα είναι στο δυνατόν πιο ουδέτερος κριτής, που ταυτόχρονα όμως θα κάνει σεβαστή και την ομοθεσία του κράτους. Και έτσι, αν υπήρχαν σωστέ προσφυγέ με κάποιο δημοσιολαβητή, δεν θα χρειαζόταν να εμπλεκόμαστε εμεί ε, ε, στα εσωτερικά και στην νομοθεσία των κρατών αυτών. Με έκπληξη βλέπω ότι υπάρχει μια αναφορά σε. μόνο μία αναφορά σε διαμεσολαβητή από μια από τι αναφερόμενε που μίλησε για απόρριψη τη πρόταση για εξέταση τη δική τη αναφορά από τον Εθνικό Διαμεσολαβητή τη Δανία. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν φαίνεται ασχοληθεί. Πάντω είναι θέματα πάνω απ' όλα και Ευρωπαίου βεβαίω διαμεσολαβητή, αλλά και του δικτύου που αναπτύσσει με του εθνικού διαμεσολαβητέ. Και εάν ένα διαμεσολαβητή δεν επιτελεί το καθήκον του, θα πρέπει να καλείται από τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή να φροντίσει να επιλύσει αυτά τα ζητήματα. Και αυτά βεβαίως είναι ίσως η πιο ήπια μέθοδος για να προσφέρουμε αρρωγή στον Ευρωπαίο πολίτη. Και τελευταία παρατήρηση. Με τόσες απογοητεύσεις που έχουμε ζήσει στον τομέα αυτό, νομίζω ότι πρέπει εμείς, ευρωβουλευτές κυρίως, να, μια και μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ε, πρέπει να ε, βγάλουμε το θέμα στα μέσα μαζικής και τα ΜΜΕ σε κάθε χρόνο, πιστεύω, και κράτος πιστεύω, και αυτό είναι και δικό μου τουλάχιστον δική μου ε, εντύπωση μπορούν να μας βοηθήσουν στον αγώνα για την ευαισθητοποίηση έναν ενό κρατου μέλου, το οποίο δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ λυπηρό αλλά και πολύ σοβαρό το θέμα. Σας καλώ όμω, σας εκλυπαρώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Και κύριε Γιάρ, εσεί πρώτο να είστε και πιο σύντομο. Α, όχι κυρία Άουκεν. Κοιτάξτε, επειδή είναι θέμα που αφορά την Δανέζικη Δημόσια Διοίκηση, θέλω να είναι σαφή αυτά που θα πω. Ένα ερώτημα στον κύριο Μπουλάν. Συμφωνώ με αυτά που είπε, αλλά να ξέρετε ότι ο όρος διαμεσολαβητής και ο όρος ombudsman δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στα γαλλικά, ναι, στη Γαλλία ο ombudsman είναι διαμεσολαβητής, αλλά στη Δανία άλλο είναι ο διαμεσολαβητής, δεν είναι σαν τον ombudsman. Ακούσαμε τις μαρτυρίες που μας συγκίνησαν όλους, συμφωνούμε. Και οι συνάδελφοι εδώ και εγώ έχουμε ξανακούσει τέτοιες υποθέσεις. Ως η αίρια που ήμουν και εγώ είχα ακούσει τέτοιες περιπτώσεις αλλά είναι διαφορετική αυτή τη φορά η περίπτωση. Το θέμα δεν είναι εδώ να μιλήσουμε για τον διαμεσολαβητή με τον νόμο που έδωσε ο κύριος Μπουλάν. Δεν είναι δική μας δουλειά οι συνεννοήσεις μεταξύ πολιτών ή συμπολιτών για αλληλοκατανόηση. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν εσύ έχεις δίκιο, εσύ έχεις άδικο δεν μπορούμε να αποφασίσουμε σαν να είναι θέμα ευρωπαϊκού ασύλου ας πούμε. Αυτό που είναι άδικο είναι ότι για τους αναφέροντες εννοώ, είναι ότι εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν και μπόρεσαν να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, ενώ η άλλη πλευρά δεν είχε τέτοιο δικαίωμα. Ίσως ένα άλλο λάθος είναι ότι είπαμε στους αναφέροντες αυτούς ότι το να έρθουν εδώ θα άλλαζε την κατάστασή τους έστω και για μία κεραία. Ίσως η Δανία να είναι πιο αυστηρή από άλλες χώρες ή να είναι χειρότερη κατάσταση ως προς τα παιδιά. Ακούσαμε και περιπτώσεις για τη Jugendamt. Υπάρχουν τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις και αλλού. Υπάρχουν πάντα ελλείψεις της δημόσιας διοίκησης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά το θέμα δεν μπορούμε μόνο να το αναφέρουμε σαν θέμα λαθών της δημόσιας διοίκησης γιατί δεν θα το λύσουμε εδώ. Αυτό ήθελα να το πω. Εγώ είμαι πάντοτε ταχμένη υπέρ του να σταματήσει η δανεία αυτές τις εξαιρέσεις που ζητάει πάντοτε γιατί έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και ελπίζω να το κάνει κάποτε, να το, την πείσουμε τη Δανία. Οι άλλες χώρες μέλη βέβαια έχουν άλλες συμφωνίες και δεν είναι πάντα δικό μας και μόνο το λάθος. Θα μπορούσαμε η εξαίρεση αυτή το opt-out να μην την είχαμε ζητήσει. Γι' αυτό φταίμε, ναι. Αλλά Ξέρω ότι το θέμα είναι δύσκολο και συγκινητικό, αλλά θα ήθελα να ακουστεί και η άλλη πλευρά, διότι έχετε έρθει σε επαφή με την άλλη πλευρά. Και εκείνοι έχουν δικαίωμα να εκφραστούν. Ακούσαμε οι πατέρες και μητέρες να κλαίνε, αλλά στη Δανία έχει συζητηθεί επίσης το θέμα του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία μας δίνει υπερβολικά δικαιώματα στους γονείς σε σύγκριση με τα παιδιά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι οι μισές τουλάχιστον περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν εδώ ε, δείχνουν ότι οι αρχές δεν έκαναν τίποτα. Και αυτό φυσικά Γι' αυτό λυπάμαι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ την Κομισιόν που παρουσίασε τις απόψεις της για αυτές τις περιπτώσεις, αλλά λυπάμαι επίσης και γιατί ορισμένοι συνάδελφοι είπαν πράγματα που δεν έπρεπε να πούν. Ευχαριστούμε κυρία Χάουκεν. Δεν ξέρω, ίσως η μη εδώ. Ο κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. αποφεύγουν μέλλον. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι έχουν ε, περιγράψει πολύ καλά την κατάσταση. Έχω δει και εγώ στην ακρόαση με τις επαφές που είχα και με τους αναφερόμενους γιατί θα θυμάστε ότι είχαμε προβλέψει δύο ώρες και κάτσε μέχρι τα μεσάνυχτα μαζί και με τους διερμηνείς. Γιατί αυτά που μας λέγανε δεν μπορούσε κανείς να τα αντέξει. Ήτανε, ήτανε τόσο τραγικά που δεν ήταν δυνατό να τους διακόψουμε και να σταματήσουμε τη συνάντηση. Ήταν κάτι που έπρεπε να αντέξουμε και να συστήσουμε και συναισθηματικά επίσης. Πάντως θα ήθελα να πω τώρα για την προκείμενη περίπτωση και τη Δανία. Πάρα πολύ ωραία χώρα, ωραίο τοπίο και όλα αυτά. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μάλλον κάτι σύπεται στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Και νομίζω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτά που μας λέει ότι θα, θα εκδώσει κατευθυντηρίες γραμμές για δικαιώματα, επιμέλειες, επίσκεψης, επαφής κτλ. Είναι βασικά ζητήματα του ευρωπαϊκού δικαίου. Και ναι, θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια, αλλά η ευρωπαϊκή ηθαγένεια σημαίνει ότι κανείς παντρεύεται, κάνει παιδιά, χωρίζει ενδεχομένω. Και άρα αυτό συνεπάγεται κάποιους κανόνας. Και γι' αυτό πρέπει να ρυθμιστεί και το θέμα της επικοινωνίας με τα παιδιά. Η Επιτροπή μας λέει ότι έχουν όλα ρυθμιστεί. Υπάρχει αρχή της επικουρικότητας και έχει κλείσει το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να το αφήσουμε εκεί. Πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα. Δεν αρκεί να έχει αυτό το opt-out η Δανία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ε, επιτρέπουμε διακρίσεις βάρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο όνομα της ελευθερίας ενός κράτους για opt-out. Επίσης για την Επιτροπή που δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με το θέμα αυτό, έχω την εξή ερώτηση γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτό το opt-out εγώ έχω την προσωπική αυτή εντύπωση ότι η Δανία παίρνει αυτό το opt-out ε, προκειμένου να προστατευτεί και ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί το ασύστησαμε και μετά στο fact-finding mission τι είδου ε, πρόθεση για συνεργασία ήταν αυτή. Γιατί μας προβάλλανε το, τον αυτοαποκλεισμό και μας λέγανε «Μα τι θέλετε, αφού έχουμε εμείς ε, το opt-out». Ε, μας φάνηκε ότι αυτό ακριβώ ήταν το επιδιωκόμενο, αλλά πέραν του opt-out υπάρχει και το διεθνέ δίκαιο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τη Δανία αν κάνει σεβαστό το διεθνέ δίκαιο. Γιατί αν κάνει σεβαστό το διεθνέ δίκαιο, πώ είναι δυνατόν να μη σέβεται το ευρωπαϊκό. Πώ είναι δυνατόν δηλαδή με άλλε χώρε να ρυθμίζουν τα προβλήματα, αλλά σε μια διαφορά μεταξύ Δανία και Αυστρία να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το δίκαιο, το ευρωπαϊκό, με τον αυτό το αποκλεισμό. Εάν είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει το δικαίωμα της επιμέλειας και της επικοινωνίας των ε, παιδιών, ε, να χάνει ένας ε, γονιός το δικαίωμα να βλέπει τα παιδιά του μόνο και μόνο γιατί έχει βγει εκτός της χώρας, τι κάνουμε. Και τώρα θα ήθελα, γιατί και ο Βίκτορ πολύ ωραία το περιέγραψε, να πέραν αυτών όλων που έχουμε πει, να δω τι είδους συγκεκριμένη απάντηση μπορούμε να δώσουμε στους αναφερόμενους. Γιατί πάντα βλέπουμε τις ίδιες παραβιάσεις. <laughs> θα μπορούσαμε να αποστείλουμε μια ε, να τους δώσουμε την ιδέα ότι μπορούν να απευθυνθούν στο Ευρωπαϊκό Δικοστήριο έστω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, το επικοινωνήσουμε το θέμα, να το προβάλλουμε επικοινωνιακά. Είναι ενδιαφέρον να συζητούνται στα μασομαστικής ενημερώσεις αυτά τα πράγματα που πάνε στραβά. Και επίσης η Επιτροπή θα ήταν καλό παρακαλώ να εξετάσει εάν είναι δυνατόν το opt-out να οδηγεί σε διάκριση εις βάρος πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι τελικά οδηγείται ανταψούρτουμε όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούμε με το, με το opt-out να αποκλειόμαστε, να αυτοαποκλειόμαστε από κάθε δυνατή, ε, δυνατό έλεγχο. Δεν σημαίνει απόλυτη ελευθερία το opt-out, δεν σημαίνει πάνω απ' όλα ελευθερία για διακρίσει ει βάρο των Ευρωπαίων πολιτών. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και το τελευταίο και πιο σημαντικό, τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτά δεν πρέπει να παραβιάζονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γιάρη. Η κυρία Ζητάνοκα, παρακαλώ. Θα είμαι πραγματικά σύντομη κύριε Πρόεδρε. Με όλη την κατανόησή μου προς τους αναφερμένους θα ήθελα να προβληματιστούμε τι να κάνουμε και πώς να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη την επικουρικότητα. του με τον κύριο Γιάρα ότι δεν πρέπει να μείνουμε στα βρωμένα χέρια πάντως μια που έχουμε και την ε, Επιτροπή εδώ, θέλω να πω ότι πολλές φορές ε, τα παρατάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσείς είστε ο ενδιάμερος μεταξύ των αναφερομένου, μεταξύ των πάντων της Επιτροπής Αναφορών και των, των κρατών. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις διαπιστώνεται ότι απευθύνεται η Επιτροπή προς τις κυβερνητικές ε, ακολουθεί μια τυπική απάντηση, α, τι ωραία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν ε, επιμένετε στο να σας δώσουν κάποια ουσιαστική απάντηση κυβερνικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένη. Συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις συγκεκριμένες παραβάσεις που καταγγέλλονται. Είναι απλουστευτικέ αυτέ οι απαντήσει που είναι οι κυβερνητικέ αρχέ και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένε υποθέσει και κατηγορίε. Νομίζω ότι μια που είστε εδώ πρέπει να σας πούμε, να επιμένετε, να εμένετε. Οτι αυτός είναι ο λόγος ύπαρξη της Επιτροπής των Αναφορών. Θέλουμε να μας σέβονται. Γι' αυτό υπάρχουν τα κοινωνικά θεσμικά όργανα. Δεν ανακατεύονται στα ιστορικά τους. Πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε παρακαλώ να επιμένετε περισσότερο και να ζητείτε ουσιαστικές απαντήσεις. Αυτό θα βοηθήσει τέτοιες υποθέσεις. Ευχαριστώ κύριο Μπέκερ. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμοι αναφερόμενοι, αναφερόμενες, είστε με πολύ σύντομος. Έχουμε εδώ, δεδομένη αυτή της τόσο τραγική, συναισθηματικά φορτισμένη, αλλά και πολιτική κατάσταση, ένα ζήτημα νομοθετικό, ένα ζήτημα επικουρικότητας, ένα ζήτημα opt-out. Όλα αυτά πρέπει να τα, πρέπει να τα διαχωρίσουμε, πρέπει να τα προσδιορίσουμε. Και από όλες τις προτάσεις οι οποίες διατυπώθηκαν εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε ότι πρέπει να στραφούμε προ την πολιτική πίεση, προς την πίεση από μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτό πρέπει να είναι το πρώτο στο οποίο θα καταλήξουμε, το πρώτο μέτρα και υποστηρίζω απολύτως να συνεχίσουμε και με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Να αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο έτσι ώστε να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Εκεί όμως θέλω να ξέρω και να περιμένω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να ασκήσουν πολιτική και νομική, νομοθετική δημιουργικότητα για να μας επιτρέψουν να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση αυτή, να μας λένε έτσι έχουν τα πράγματα και να είμαστε ευχαριστημένοι. Εδώ όταν έχουμε να κάνουμε δικαιώματα παιδιών λίγουν και οι ανοχές μας. Σταματάμε να είμαστε ανεκτικοί και γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε αμέσως τα ζητήματα της αλλαγής του opt-out, θα το πω, να, γίνει, να γίνουν πρώτα θέματα προτεραιότητα από πλευράς Επιτροπής και Συμβουλίου. Αυτό περιμένω να μου πούνε και να μην μου λένε έτσι έχουν τα πράγματα. Save of the same. Κύριε Βέρτμαν. Θα ξεκινήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς η απάντησή σας δεν είναι απάντηση δεν μας διαφωτίσατε καθόλου σε σχέση με αυτούς τους άντρες, τις γυναίκες, τα παιδιά. Νομίζετε ότι αυτή, αυτό το opt ότι αυτό η αυτοεξαίρεση είναι η απάντηση. Νομίζω ότι είμαστε τόσο αφελείς που να μην γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διεθνείς συνθήκες όπως η σύμβαση της Χάγης. Γνωρίζω μία ή δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είχαμε εφαρμογή της ε, Σύμβασης της Χάγης κατήσχησε το opt Μα τι είναι αυτό. Είναι αυτό Ευρώπη. Ερωτώ κυρίες και κύριοι. Συχνότερη συνεργασία λέτε. Μα εγώ έχω πάρα πολύ ε, κοντινή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ στενή συνεργασία για μια σειρά αναφερομένων. Και δυστυχώς απάντηση ήταν μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε και όχι παραπέρα λόγω του opt-out. Εγώ να σα πω την αλήθεια το αμφισβητώ. Δεν νομίζω ότι κατησχεί το opt-out του, του, του, επί του θεμελιώδη χάρτη των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Δεν κατησχεί κανένα άλλο ευρωπαϊκού δικαιώματο. Μιλάμε εδώ, αγαπητοί μου, για μια ευρωπαϊκή χώρα, μια χώρα που αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνοι, εντάξει, υπάρχει το opt-out, αλλά δικαιούται επί τη βάση αυτού το συγκεκριμένο κράτος να λέει όχι στην εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου, να λέει όχι στα ευρωπαϊκά, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην είναι το να δεχόμαστε κάτι τέτοιο Μάργαρετ, γελά, σε βλέπω το, το, το Όμως, ε, βλέπουμε τη ζωή και άκρα αριστερά και άκρα δεξιά τέτοιε τάσει, αλλά το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να κρατήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη θέση του, αν μπορούμε να φροντίσουμε του ε, νεαρού Ευρωπαίου, ε, του, του, τους αναφερόμενους. Μα αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε ε, είναι εδώ να, να, να μείνει όρθια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλος ανέφερε τους Εβραίους, άλλος τους Ναζί και καθόμαστε και ακούμε τέτοια πράγματα από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μα είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τέτοια πράγματα. Είμαστε πολιτικοί. Έχουμε αυτά τα δικαιώματα εδώ που θίγονται των αναφερομένων των συμπατριωτών μας. Συμπατριωτών γιατί ζούμε όλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το να επιτρέψουμε να ποδοπατιούνται έτσι αυτά τα τρώνε δικαιώματα, να τα πετάμε στα σκουπίδια τι του, του, τα παιδιά τους. Όχι, όχι, σε παρακαλώ, Έχουν το δικαίωμα τα παιδιά να είναι με τη μάνα τους. Η μάνα τους τα γέννησε. Οπότε, σας ερωτώ. Οι μανάδες και οι πατεράδες σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υφίσταται τέτοια μεταχείριση. Μπα και η Δανία μεταχείριζεται καλύτερα τα ζώα από του ανθρώπους. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σας πω. Α, έχω μια σειρά θεμάτων να θίξω. Έχουμε προβλήματα με τις ε, αρχές. Σκεφτείτε τι γίνεται με τα έγγραφα. Σε μια δύο περιπτώσει που σήμερα εξετάσαμε, έχουμε περιπτώσει κατά τι οποίε έχουμε λάθο όσον αφορά τα έγγραφα. Κάποια κυρία μπορεί να αποδείξει ότι είχε ένα γραφό στα χέρια της, αλλά κάποια στιγμή εκδόθηκε άλλο εγγραφό, το οποίο όμως ήταν ευμενές για τον πρώην σύντροφό της. Άλλες φορές τους αρνούνται την πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα. Έχει να κάνει αυτό με το opt-out, ή είναι αυτό ευρωπαϊκό δικαίωμα. Μια φορά κάποια στιγμή πήραν τηλέφωνο. Κάποια κυρία, κάποια αναφερόμενη, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε να την συμβουλεύσω. Τι να κάνει. Εξαφανίστηκαν τα έγγραφα. Δεν υπάρχουν πλέον αποδείξει. Να τον επιτρέπουμε τέτοια πράγματα. Τι λέτε εσείς από την Κομισιόν. Για να ρωτήσουν τι γίνεται στα κράτη-μέλη. Τι είναι αυτό. Είναι αυτό Ευρώπη. Αμφιβάλλω εντόνως. Κάτι άλλο τρόπο θέλω να σας πω. Πρέπει να σας το πω. Φυλακίζονται τα παιδιά μας. Τα ακούσαμε σήμερα. Τα ακούσαμε και στην αποστολή στη Δανία. Τα παιδιά δεν μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Δανίας. θέλουν να πάει δύο μέρες ή λίγες εβδομάδες μια μάνα και δεν την αφήνουν να πάει διακοπές με το παιδί της. Πρέπει να μείνει στη Δανία. Μα είναι δυνατόν να μην αφήνουν τα παιδιά να βγουν έξω από τη χώρα να δουν κάτι άλλο. Θέλουμε τέτοιο πράγμα για τα παιδιά μας. Επίσης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μεσολαβητής. Τον έχουμε δει, τον έχουμε συναντήσει. Και τι μα είπε, συνάδελφε. μα είπε το τι μπορεί να κάνει η υπηρεσία του. Σήμερα ακούσαμε τι είπε σε μια αναφερόμενη. Ε, είναι δυνατόν να συνομιλούμε με τον δημοσιολογητή όταν έχουμε τέτοια αντιμετώπιση. Κάτι άλλο τώρα. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα ίδια. Αλλά πρόκειται για ένα πάγιο πρόβλημα στην Δανία. Εντάξει. Και σε άλλες χώρες υπάρχουν προβλήματα φυσικά. Εδώ όμως το πρόβλημα αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Είναι, ε, είναι κάτι που προκύπτει συνέχεια. Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μιλάμε για πολλέ εκατοντάδες τέτοιων υποθέσεων. Άρα όλα μαζί κάνουν χίλιες περιπτώσεις τέτοιες. Τι είναι αυτό, είναι φυσιολογικό, είναι ευρωπαϊκό, είναι εντάξει να, έχουμε μια τέτοια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγχαρητήρια στους αναφερομένους. Συγχαρητήρια για το θάρρος τους που ήρθαν εδώ, που ήρθαν και, το, τα βγάλανε στη φόρα, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ενήμερη σε σχέση με το τι συμβαίνει. Σε ένα κράτο μέλος το οποίο απολάβει τόσες εκτιμήσεις. Εγώ τρέφω πολλές αμφιβολίε για το κατά πόσον είναι δυνατόν αυτή η γνώμη για την Δανία να συνεχίζει να ίσχυει. Εντάξει, σας άκουσα. Πολύ ωραία αυτά που μα είπατε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά για σκεφτείτε τα. Γιατί σύντομα δεν θα έχουμε μεικτά ζευγάρια. Γιατί, γιατί πριν από λίγες μέρες, τι άκουσα στη Γερμανία, στην Αυστρία. Θα παντρευτώ μόνο Αυστριακό ή Αυστριακή γιατί δεν θέλω να, να πάθω αυτά τα οποία άκουσα να συμβαίνουν όπως άκουσα στο κοινοβούλιο. Να, αυτό, αυτό άκουσα από κάποιο νέο. Και καταλαβαίνω γιατί το σκέφτεται. Συμφωνούμε νομίζω τελικά ότι αυτό θα πρέπει να κατέβει στην Ολομέλεια. Τα είχαμε ξαναπεί και πριν από δύο χρόνια. Αλλά ποια ήταν η αντιμετώπιση. αυτό είναι συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι αυτά τα προβλήματα όχι, δεν είναι συγκεκριμένες, εξατομικευμένες περιπτώσεις. Ούτε απλές περιπτώσεις. Επομένως, ας έχουμε αυτό κατά νου. Τόσες λεπτομέρειες έχουμε Α, κάτι άλλο. Αγαπητή κύριε Επιτροπή, υπήρξε κάτι το οποίο διαστρεβλώθηκε. Ήταν αυτή η υπόθεση του, του Αυστριακού, της Αυστριακής. Δεν ήταν εκείνη ο απαγωγιας η η απαγωγιας Διαστρεβλώθηκε. Γιατί διάβασα τη δήλωση ε, και όπως διορθώθηκε ε, που διαβάστηκε στην κυρία Ματσόνη. Πρόκειται για τα του Κοινοβουλίου. Αυτά τα οποία εμείς τα λαμβάνουμε από τους αναφερομένους. Και δεν είναι απλώ. γνώμη, πρόκειται για τεκμήρια. Και αυτό θα πρέπει να το ψάξουν. Τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, σα το επισημαίνω. Επισημαίνω σε όλου ότι οι ευρωβουλευτέ μπορούν να αποφανθούν μόνο επί τη βάση των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους, από ό,τι τους δώσανε και από ό,τι ερεύνησαν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ορισμένοι αμφισβητούν την αξιοπιστία μας. Το έργο μας. Σύμφωνοι, δεν είμαστε δικαστήριο, αλλά δεσμευόμεθα από το καθήκον μας ως μέλη της Επιτροπής των Αναφορών. Θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό τους για να πετύχουν κάτι. Ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε πίσω τα παιδιά τους. Να ξαναβρούν λέει τα παιδιά τους οι μανάδες και οι πατεράδες αυτοί. Σας ευχαριστώ όλους. Πολύ σοκαριστικό το πρωινό. Μήπως θέλετε να προσθέσετε τίποτα κύριε Μποστινάρο. Θα κάνω συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, προφορική ερώτηση με συζήτηση και ψήφισμα. Δύο, Επιστολή προς τον Κομισιόν για να αρχίσει να επεξεργάζεται ένα έγγραφο για το πρόβλημα σε πανενωσιακό επίπεδο. Έχει σημασία και η συγκεκριμένη χώρα, αλλά συμβαίνουν και σε άλλες. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, να ζητήσουμε από την Κομισιόν να καταλήξει σε μία νομικά δεσμευτική λύση για να αποτραπούν τέτοιες τραγωδίες. Κύριε Μποστινάρο, και εγώ θα έλεγα κάτι τέτοιο, γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Προέδρου. Μου τον παίρνετε. Λοιπόν, καταλήγω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν σοκαριστικό το πρωινό. Με θύμισε τον Σέξπιρ που είπε «Something is wrong in the kingdom of Denmark». Ω, δεν τελείωσα, περιμένετε. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Είναι ιδεολογικό. Και έχω σοκαριστεί γιατί συμβαίνει σε μια χώρα στο βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. It's very strongly. Και νομίζω ότι πλήττει γενικά την ευρωπαϊκή ιδέα. Αναρωτιέμαι τι κάνουν οι Δανείοι βουλευτές για να αλλάξουν την κατάσταση. Αλλά δεν είναι δικό μου θέμα αυτό. Η κυρία Χάουκεν θα ήθελα να κάνει μια προσπάθεια να τους πληροφορήσει εκεί στη Δανία, στη Δανέζικη Βουλή. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Μπορούμε να γράψουμε και άλλη επιστολή προς τις Δανέζικες αρχές ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα απαντήσουν πιο συγκεκριμένα. Όχι λέτε εσείς. Ο Δαβίδ λέει να το κάνουμε. Βέβαια πρέπει να γνωρίζει και ο Επίτροπος ακριβώς τι συμβαίνει με αυτές τις αναφορές και τα υπόλοιπα. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της κατάθεσης ερώτησης στο Κοινοβούλιο και συζήτησης. Αυτό όμως θα αποφασιστεί στη, στους συντονιστές. Έληξε, όχι, όχι, πρέπει να σας πω ότι η δανέζικη κυβέρνηση έχει απαντήσει επανειλημμένος Μπορεί να μην σας ικανοποιούν οι απαντήσεις, το ξέρω αυτό, αλλά έχει απαντήσει. Κρίμα που πρέπει να τελειώσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ τους αναφέροντες και τους συναδέλφους. Ελπίζω η Κομισιόν να καταλήξει σε κάποιες δυνατότητες βοήθειας προς τις περιπτώσεις αυτές και θα τη στηρίξει και το Κοινοβούλιο. Η επόμενη συνεδρίαση. Α, όχι, το τελευταίο θέμα ήταν αν θα κρατήσουμε ανοιχτές ορισμένες περιπτώσεις. 45 και 47 θα μείνουν ανοιχτές. Στο